Good afternoon. Καλησπέρα σας. Καταρχήν ε, η πρόεδρος θα καθυστερήσει λίγο, αλλά θα αρχίσουμε εγκρίνοντας καταρχήν την ημερήσια διάταξη. Μετά από αίτημα τελευταία στιγμής της διάσκεψης των Προέδρων, Προσθέτσαμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον Ζαν Λουί Μπορλό. Θα προσθεθεί λοιπόν αυτό το θέμα στην αρχή της συνεδρίασης, έτσι αποφασίστηκε. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο μυρίσιας διάταξης με αυτή την προσθήκη για την ανταλλαγή απόψεων. Ναι. Εγκρίνεται. Τώρα οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης όπως ξέρετε τελειώνει με μια εκδήλωση στο Λουξεμβούργο στις 9 Δεκεμβρίου όπου θα πάνε οι Υπουργοί Ανάπτυξης των χωρών μελών, η Φρυδερίκα Μογκερίνη και εκλήθηκε η πρόεδρος μας και τα τρία όργανα θα συνυπογράψουν και κοινή δήλωση. Στην επόμενη Ολομέλεια, στις 2 Δεκεμβρίου, θα τα πούμε και εκεί, θα ανακοινωθεί και εκεί. Επίσης την Τετάρτη θα υπάρχει προφορική ερώτηση. Was, uh, our question from this committee. Ένα πρόσθετο θέμα και τέλος Στο τέλος της αυριανής μας συνεδρίασης ο Επίτροπος Στυλιανίδης uh, uh, θα μιλήσει για την κρίση των Δημητριακών. Τώρα τα πρακτικά 14 Ιουλίου και 8 Οκτωβρίου είναι στους φακέλους σας αν έχετε κανένα σχόλιο παρακαλώ να πληροφορήσετε σχετικό στη γραμματεία πριν λήξει η σημερινή συνεδρίαση και αλλιώς θα εγκριθούν. Τέταρτον, έγκριση των αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών της 10ης Νοεμβρίου και αυτά στους φακέλους σας. Αν έχετε σχόλια να το πείτε στη γραμματεία πριν λήξει η σημερινή συνεδρίαση και ακόμη μια φορά εάν δεν ληφθούν σχόλια θα εγκριθούν και αυτά. Πέμπτον, ανακοινώσεις της Καμισιόν. Έχει καμία ανακοίνωση η Καμισιόν? Όχι, όχι. Το καινούργιο λοιπόν θέμα που προσθέθηκε η ανταλλαγή απόψεων με τον Ζαν Λουι Μπορλό, ηγέτη της οργάνωσης Ενεργή Πουρλαφρίκ. Όπως ξέρετε η πρόσβαση στο, στην ηλεκτρική ενέργεια είναι βασική για την ανάπτυξη και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα και πλαίσια όπως η βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ Ξέρετε ότι η ενέργεια είναι πολύ σημαντικό καθώς και το εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. που είναι θέμα που και εμείς το προσέχουμε ιδιαίτερα Χαιρόμαστε λοιπόν που έχουμε μαζί μας τον Ζαν Λουί Μπορλό Έχουμε ακούσει για αυτή την Ολομέλεια, είχαμε ακούσει στην προηγούμενη Ολομέλεια, αλλά μάλλον τα μέλη θα θέλουν κάποιες περισσότερες πληροφορίε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Μπορλό που προσήλθατε σήμερα. Ξέρω ότι είναι πολύ επίκαιρη η συνάντησή μας σήμερα γιατί αρχίζει και η διάσκεψη των Παρισίων. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί παλαιοί συνάδελφοι, ε, γιατί πρέπει να σας αποκαλέσω έτσι, γιατί είχα την τιμή να είμαι μέλος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ την πρόεδρο κυρία Λίντα Μακάβανη, η οποία είχε ε, δεχτεί αυτήν την συζήτηση στη διάσκεψη των ε, πρόεδρων των ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα θέμα ε, το οποίο μπορούμε πλέον νομίζω να δούμε με πιο άμεσο και επιχειρησιακό τρόπο. 14 χιλιόμετρα από την Ευρώπη υπάρχει μια Ήπειρος ε, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο αναβρασμό. Ε, θετικό αναβρασμό αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνο. 14 χιλιόμετρα λοιπόν τα για μία Ήπειρο ε, η οποία ήταν 185 εκατομμύρια τον προηγούμενο αιώνα και έφτασε στο 1 ε, δις τώρα και προχωράει ε, χωρίς επιστροφής για να φτάσει στα 2 δις και κάτι. Δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της Αφρικανικής Υπήρου, στην, της οποίας 50% του πληθυσμού δεν είναι, είναι κάτω από 20 ετών, ε, είναι ότι έχει υπάρξει αντικείμενο ε, της μεγαλύτερης ηλεκτροδότησης του κόσμου. Τα πρότυπα ε, τα οποία έχουν προχωρήσει τώρα είναι συγκεκριμένα αλλά από τα 980 εκατομμύρια ε, σε όλη την Ιφίλιο που δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό, τα 700 ζουν στην Αφρική. Ε, τρίτο στοιχείο, ε, πριν από μερικά χρόνια στις δεσμεύσεις ας πούμε της χιλιετίας ε, η δέσμευση για την ενέργεια ήταν ένα μικρό υπόμνημα ενώ τώρα και μια μικρή αναφορά ενώ τώρα θεωρείται ε, ε, δικαίωμα γιατί ταυτόχρονα με την πρόσβαση στην ενέργεια έχουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στο ηλεκτρισμό, πρόσβαση στην ελευθερία, στη χειραφέτηση των γυναικών, στην κοινωνική ζωή και πολλά άλλα. Όταν τα τρία τέτοια μια ε, μιας υπήρου δεν έχει φως. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλές λέξεις, ε, αναπόφευκτα μαζικά προχωρούν προς τα σημεία τα φωτισμένα, τα, τις πρωτεύουσες δηλαδή στην Αφρική, τα μεγάλα λιμάνια κτλ. Αλλά φυσικά έχει ξεκινήσει ήδη η ε, μεγάλη πορεία των ανθρώπων και δεν θα μιλάμε πλέον για τα πολύ λίγα εκατομμύρια σύρων, αλλά θα μιλάμε για ε, ε, κάτι τελείως διαφορετικό. 800, εκατομμύρια κινητά πουλήθηκαν μέσα σε 8 χρόνια στην Ήπειρο αυτή. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ε, να πούμε ότι δεν θα προχωρήσει προς την ε, προς το φως. Όταν 25% της ηλεκτροδότησης ε, ε, αναπτύσσει την, αυξάνει την ανάπτυξη κατά 5% και όταν όλοι οι οικονομολόγοι καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιο πλουτισμό. Η Αφρική είναι ο πιο κοντινός μας εταίρος. Είναι ο εταίρος μας για την ανάπτυξη τώρα που βρίσκεται σε στάσιμη ε, κατάσταση ο εταίρος της ε, Ασίας και ε, ε, οπωσδήποτε θα πρέπει και οι, οι μεσαίες να είναι αυτές στις οποίες θα απευθυνθούμε για την ανάπτυξη αυτή. Όλα λοιπόν εξαρτώνται από την ενέργεια και επομένως εδώ δεν μιλάμε απλά για μία προτεραιότητα. Για προσωπικούς λόγους ε, για λόγους υγείας μάλλον εγκατέλειψα τη δημόσια ζωή για κάποια διάστημα, για κάποιο διάστημα, για κάποια χρόνια ε, και κάποια στιγμή το 2008-2009 ήταν σε επαφή μαζί μου ή ε, κάποιοι ηγέτες Αφρικανοί που μου είπαν άκουσε Ζανλουί δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Προσπάθησε να κάνεις μια διάγνωση, προσπάθησε να μας κάνεις μια πρόταση κυρίως εν ώψη των μεγάλων των μεγάλων γεγονότων και ακρο... Ε, σημαντικών γεγονότων, ένα εκ των οποίων ξεκίνησε σήμερα το πρωί και γι' αυτό ζήτησα να έρθω το απόγευμα, γιατί ήθελα να ε, είμαι ε, παρόν και βεβαίως ε, θέλουμε αυτήν την, ε, ε, την δημόσια πούμε παρέμβαση για να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια να επιτύχει αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Και ο δεύτερος λόγος, ο πουθενά μαζικό ε, πρόγραμμα ηλεκτροδότησης, ε, όχι απλής χρηματοδότησης, ε, αλλά πουθενά και ποτέ στον κόσμο, ούτε καν τη δεκαετία του 30, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στο Βέλγιο. Ποτέ, μα ποτέ δεν υπήρξε μαζικό πρόγραμμα χωρίς ένα τμήμα δημόσιας ε, χρηματοδότησης για τα πιο περίπλοκα, για τα πιο ε, απομακρυσμένα σημεία, για την εξασφάλιση της φερενγιότητας του προγράμματος κτλ ο Jean-Claude Juncker, ο François Hollande είχαν πει ότι εμείς θα θέλαμε ένα πραγματικό σχέδιο με την ε, Αφρική. Θέλουμε να συμφωνήσουν όλοι όσο γίνεται περισσότεροι με μια πραγματική διακυβέρνηση. Και στις 15 Ιουνίου του 2015 ελήφθη η απόφαση. Η ε, ε, η επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής ε, ε, ε, σε συνεργασία και ενώπιον του Κοινοβουλίου των Λαών της Αφρικής, αντίστοιχο με το δικό σας. Όλοι αυτοί επιθυμούν να έχουν ε, συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα αυτό είναι και το πρώτο μήνυμα που θέλω να σας ε, μεταφέρω κύριε Πρόεδρε. Από την άποψή μου είναι ζωτική σημασία στα δύο κοινοβούλια αυτά να μιλούν, να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν επισκέψεις ε, γιατί είναι σημαντικά για μας αυτά που γίνονται στην Αφρική. Δεν είναι δυνατόν, είναι πολύ επικίνδυνο μάλιστα να μην τα θεωρούμε σημαντικά. Ε, ωραία, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτήν την ε, παναφρικανική εταιρεία, αλλά εσείς, ε, εσείς σαν Ευρωπαίοι θα μας βοηθήσετε. Η ευρωπαϊκή πλευρά είναι έτοιμη για, σε όρους ειρήνης, σε όρους σταθερότητας, σε όρους ηθικής βοήθειας, σε όρους συνοχής ενός μεγάλου project, ενός μεγάλου σχεδίου Μπορεί η Ευρώπη, λέω, να αναλάβει τα ενία μαζί με ε, τους φίλους από τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, να υπάρχει ας πούμε ένας εκπρόσωπος από τους Ρεπουμπλικάνους, άλλος ένας από τους Δημοκράτες, μαζί με το Κοινοβούλιο, μαζί με την Κομισιόν, μαζί με τους Ιάπωνες Ε, πρόκειται για μία ήπειρο ε, η οποία σε λίγο θα ε, είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο να δεσμευτεί όχι οικονομικά αλλά να πει ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους λαούς της Ευρώπης θεωρούμε ότι είναι στρατηγική σημασία μια σε βάθος συζήτηση και μια και βρισκόμαστε μεταξύ μας και δεν έχουμε δημοσιογράφους να σας πω ότι λυπούμε. Έχουμε εργαλεία όπως είναι ας πούμε ε, η διευκόλυνση κοτονού κτλ αλλά δεν έχουμε στρατηγική. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Και δεν είναι καλό που δεν είναι παρούσα η Κομισιόν, ας πούμε. Θα πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση και νομίζω ότι ε, μια και όλοι έχουμε τις συνήθειές μας και μια και η Κομισιόν ε, έχει αναλάβει τα καθημερινά ας πούμε, ε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να τίνει τη χείρα βοηθείας, ε, να πει το Κοινοβούλιο και να καταλάβει ότι μας περιμένει η Αφρική, στρέφεται προς εμάς. Η Αφρική έχει αυτό το παράδοξο ότι έχει το μεγαλύτερο δυναμικό ε, για τη, στην γεωθερμία, στην, ε, στον υδροηλεκτρισμό, ε, στους, στην, στη βιομάζα, στην, στη ηλιακή ενέργεια στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς επίσης και την αιωλική στην, στα ύψη της Αιθιοπίας, καθώς επίσης και στην πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού, αλλά αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει στρατηγική έτσι ώστε ε, να προχωρήσει ε, το πράγμα. Και βεβαίως ε, δεν είναι ακριβώς αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι μας ενδιαφέρει, είναι δικό μας ζήτημα τελικά αυτή η ενεργειακή προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να το κάνουμε γιατί διαφορετικά η άποψή μου η προσωπική είναι ότι αν σε, μέσα σε πέντε χρόνια ας πούμε δεν έχει κάνει κάτι η Ευρώπη τότε θα πέσουμε τελικά σε ένα κλίμα κλίμα φόβου και θα είναι πάρα πολύ κακό. Ε, ε, διαφορετικά θα αφήσουμε την Αφρική στο έλεος των, ε, ναρκο, των ναρκωτικών και των εμπόρων ναρκωτικών. Θα υπάρξει αστάθεια η οποία κάποια στιγμή ενδεχομένως θα φτάσει σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση όπου στην υποσαχάρια Αφρική τα πράγματα δεν θα, θα ξεφύγουν από τα όρια και επομένως νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχει κανένα ένα μέλλον η Αφρική. Εμεί πρέπει να βοηθήσουμε να δεσμευτούμε έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη στην Αφρική συντονισμένη και έτσι ώστε ε, η ανάπτυξη αυτή να έχει καλά αποτελέσματα και στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς. Αν υπάρχουν ερωτήματα, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία, γιατί υπάρχουν εδώ μέλη από την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά και μέλη της Μικτής κοινοβουλευτική Αντιπροσωπείας με τις χώρες ΑΚΕ. Και η συνεδρίαση της Ισομερούς Συνέλευσης θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και φυσικά τα, η θεματολογία αυτή ενδιαφέρει και τους βουλευτές από την ε, Ισομερή Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΑΚΕ και θα συζητήσουν προφανώς και αυτές τις πληροφορίες που αναφέρατε. Είναι σημαντικό λοιπόν να συζητηθεί και από τις δύο πλευρές. Ο κύριος Νόησερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπολό. Το θέμα που αναφέρατε και από και για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος ότι χωρίς την, ε, τους ενεργειακούς πόρους δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και αντίστροφα η ανάπτυξη μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη δραστηριότητά μας. Το 2012 είχα εκπονήσει μια έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την ενέργεια στις υποανάπτυξη χώρες και στην ε, έκθεση αυτή είχα τονίσει ότι είναι απαραίτητο το Κοινοβούλιο να δώσει περισσότερες χρηματοδοτήσεις, να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, ώστε και στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ίσως η Κομισιόν δεν το έχει πράξει αυτό το οποίο ζητήσαμε επαρκώς, αλλά εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή και η απόφαση του Κοινοβουλίου που ακολούθησε έδειξαν σαφώς την πολιτική μας θέληση σε ό,τι αφορά τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ενεργειακά θέματα στι αναπτυσσόμενε χώρες. Εγώ εκπλήσω με λιγάκι γιατί είπατε ότι, είπατε ότι δεν είναι θέμα ε, χρηματοδότησης αλλά είναι θέμα του μηνύματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου που πρέπει και οι δύο αυτές πλευρές να εγγύψουν στο θέμα αυτό. Γι' αυτό θέτω και το ερώτημα αυτό εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό οι ενέργειε σε αυτόν τον τομέα, γιατί υπάρχει περιθώριο στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως χρειάζεται καλύτερο συντονισμό, και εξάλλου νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο για τέτοιε ενέργειε, Αλλά αυτό το πολιτικό πλαίσιο έχει θεσπιστεί και από τα Ηνωμένα Έθνη με την πρωτοβουλία του Μπανκιμούν Ενέργεια για Όλους. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Η πρωτοβουλία της Αφρικής θα συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Θα μπορέσουν από κοινού να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ξέρω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κάνει ιδιαίτερα πολλά στον τομέα της, στον χώρο της ε, Δυτικής Αφρικής και υπάρχουν εθνικά σχέδια για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Δυτικοαφρικανική Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ε, παροχής ενεργειακών πόρων. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πώς βλέπετε εσείς προοπτικές για συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και ποια είναι και η δική σας εικόνα σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν για χρηματοδότηση στα θέματα αυτά. Κατά τα άλλα, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Χρειαζόμαστε να κάνουμε μια εργασία πυθούς, μια εργασία ε, υποστήριξη των προοπτικών της ανανεώσιμη ενέργειας για τις χώρες που είναι υπό ανάπτυξη. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Θα μπορούσε η Κομισιόν ο πρεσβευτής κύριο Ρουντόλφι να λάβει το λόγο και να μας παρουσιάσει θέση τη Κομισιόν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ και σας κύριε Μπορλό για αυτό τα εμπνευσμένα λόγια για τη σημασία της ενέργειας και τον κύριο Νόησερ επίσης. Αποδέχομαι εκ μέρους της Καμισιόν 300% αυτά που είπε ο κύριος Μπουρλό. Το 2008 ήδη, από εκεί αρχίζω, ο κύριος Τούρμες ανέλαβε μία πρωτοβουλία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα και ιδρύθηκε ένα ιδιωτικό ταμείο που λεγόταν Τζερεφ μέσω του οποίου χρηματοδοτούσαμε τις ανανεώσιμες και την αποδοτικότητα και στον ιδιωτικό τομέα. Ένα ευρώ αναφορολογούμενο για, τις, ε, για τα θέματα αυτά μαζέψαμε. Και εφαρμόστηκαν και οι λεγόμενες blending facilities έχει δίκιο ο κύριος Μπουρλό. Εδώ πρόκειται για τομέα όπου δωρεές μπορούν να είναι καταλύτες, να αποτελέσουν καταλύτες και να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου για τους επενδυτάς. Η ενέργεια βέβαια είναι οικονομικός τομέας και έτσι πρέπει να την θεωρούμε. Λοιπόν αυτές οι blending facilities μαζί με την ΕΤΕ, την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά ενίσχυσαν τις δωρεές που είχαμε μαζέψει από ιδιώτες. Το Agenda for Change μετά εφαρμόστηκε για να συνδυάσει την ενέργεια με τη γεωργία που είναι οι μόνοι δύο τομείς που, με τους οποίους ασχολείται. Ξέρω ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης έγκριση του προγράμματος αυτού από το Κοινοβούλιο, αλλά αυτή ήταν η γενική κατεύθυνση που είχε δώσει τότε το Συμβούλιο. Το 12 στις Βρυξέλλες έγινε το πρώτο βήμα και συνάντηση για τη βιώσιμη ενέργεια. Ο Μπαν Γεν Γραμ είχε έρθει και ο κύριος Βαν Ρόμπουι μαζί του κάλεσαν τους ηγέτες να μαζευτούν στις Βρυξέλλες για πρώτη φορά. Το 13 με 14 τον σχεδιασμό των προγραμμάτων του εργαλείου συνεργασίας για την αναπτυξιακή συνεργασία το συζητήσαμε με συγκεκριμένες χώρες για να δούμε ποιες θα ήθελαν να λάβουν ποιους τομείς. Από την προηγούμενη από δύο χώρες στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο τώρα έχουμε 35 χώρες που επέλεξαν την ενέργεια ως κύριο τομέα για να στοχεύσουμε στη αναπτυξιακή βοήθεια, στην Αφρική κυρίως. Το 2014 επίσης <clears throat> είχαμε πει ότι το θέμα δεν είναι μόνο η χορήγηση και κατανομή κονδυλίων αλλά και θέμα πολιτικής θέλησης. Όταν ήμουν πρέσβη στην Ουγγάντα Είχα συζητήσει με τον πρόεδρο για την ενέργεια. Μου έλεγε δεν θέλουμε φιλανθρωπία, θέλουμε γιγαβάτ. Το 14 λοιπόν έγινε η ανακοίνωση για την, τον συνδυασμό με τον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να το συνδυάσουμε. Και το 15 τελειώνω άρχισε το πρόγραμμα Electrify για την πρόσβαση στον εξηλεκτρισμό στην Ήπεθρο, στην Αφρική, όπου δεν πηγαίνει κανένα ιδιωτικό κονδύλιο μέχρι τώρα. 3,5 δισεκατομμύρια για την ενέργεια, 2,5 για την Αφρική και η πρωτοβουλία αυτή για την πρόσβαση λοιπόν έχει αναγνωριστεί και στα ΣΥΠΑ, οι οποίες μας έγραψαν μια επιστολή όπου λένε ότι θέλουν να μας δώσουν, δωρήσουν 10 εκατομμύρια δαλάρια. Ελπίζω όλοι να αναγνωρίσουν τον ηγετικό ρόλο του προγράμματος Access to Energy. Ευχαριστώ. Νομίζω καταλάβατε με μια πρώτη ματιά που βρισκόμαστε εδώ, η θέση της Κομισιόν λοιπά Όλοι καταλαβαίνουμε δηλαδή τη σημασία του θέματός σας. Το θέμα είναι πώς η πρωτοβουλία που μας εξηγήσατε μπορεί να συνδυαστεί με τις υπόλοιπες προσπάθειες της Ένωσης. Τώρα αν θέλετε σε δύο-τρία λεπτά να καταλήξετε. Ευχαριστώ λέει Μπολό. Το θέμα αυτό δεν είναι ποιος κάνει τι και τα λοιπά. Χρειάζεται πραγματικά να ανεβάσουμε ταχύτητα και να βελτιώσουμε την οργάνωση. Έχουμε ζητήσει από τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής να οργανωθούν καλύτερα και να φτιάξουν μια ομάδα υψηλού επίπεδου, όπως έγινε και με την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, για να μπορέσουν να βοηθήσουν σε όλα αυτά τα σχέδια. Είναι απαραίτητο να έχουν κάποια βοήθεια, να έχουν κάποιες σηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως θα πρέπει να συνενώσουν τις προσπάθειες όλων των δωρητών της Κομισιόν, των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Είναι κατεπήγον. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό όλα αυτά τα σχέδια να είναι λειτουργικά. Κύριε Νόιζερ, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχουν ασκήσει μια πολιτική πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση Ελπίζουμε ότι στα τέλη Ιανουαρίου, τέλη Φεβρουαρίου θα μπορέσουν όλοι αυτοί να, που ενδιαφέρονται για αυτό το, το εγχείρημα να είναι παρόντες. Αλλά εξακολουθεί να ισχύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 10 εκατομμύρια παραπάνω το κάθε χρόνο. Έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από, την, από τις αφρικανικές χώρες χωρίς τη δική μας υποστήριξη, χωρίς τη χρηματοδότηση, χωρίς τις δημόσιες αρχές και τη συμμετοχή των Αμερικανών και άλλων που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους. Εμείς λοιπόν σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Φυσικά αυτοί θα πρέπει να αποφασίσουν για τις λειτουργικές λεπτομέρειες με το δικό μας έλεγχο προφανώς. Ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες που μας δώσατε και φυσικά θα είμαστε και πάλι σε επαφή στα πλαίσια της ισομερούς συνέλευσης. Το, τώρα αγαπητοί συνάδελφοι ερχόμαστε στην εξέταση των τροπολογιών προς την ε, έκθεση πρωτοβουλίας για τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά την ΤΙΣΑ, την ε, Συμφωνία για, την, ε, για το Εμπόριο Υπηρεσιών. Ξέρω ότι είναι 69 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και υπάρχει ένα αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Λόλα, στην κυρία Λόλα Σάντσε, που είναι η συγγήτριά μα για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους τους κοιόδη συγγητές. αν ε, δούμε ποιε ήταν οι αρχικέ ε, διαφορέ απόψεων, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε σε συμβαστικέ τροπολογίε που υπογραμμίζουν τι βασικέ θέσει τη Επιτροπή μα για την ΤΙΣΑ. Αν εγκριθεί η ΤΙΣΑ, θα έχει σημαντική επίπτωση στι αναπτυσσόμενε ε, χώρε και γι' αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου δεν πρέπει να έρθει σε σύγκρουση με την πολιτική ανάπτυξη και θα πρέπει να υποστηρίξει αντίθετα του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, Είναι πάρα πολύ σημαντική και η διαφάνεια σε μια δημοκρατία. Είναι απαραίτητο να γίνονται δημόσιε οι πληροφορίε σε σχέση με τι διαπραγματεύσει τη ΤΙΖΑ και είναι απαραίτητο να ακούσουμε και την άποψη των πολιτών, των ΜΚΟ, των ε, ενώσεων τη ε, κοινωνία των πολιτών και των συνδικάτων, όχι μόνο στο βορρά, αλλά και στο νότο του πλανήτη μα. Είναι απαραίτητο να δεσμευτούμε για ενίσχυση του πολυμερού πλαισίου στα εμπορικά θέματα και από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να υπονομεύει τα φόρουμ όπου είναι όλοι εκπροσωπούμενοι με δίκαιο τρόπο, θα πρέπει να ενισχύσει αυτά τα φόρα. Είναι απαραίτητο στα πλαίσια τη βιώσιμη ανάπτυξη τα κράτη να έχουν τη δική του αυτονομία για να μπορούν να εφαρμόσουν πολιτικέ οι οποίε εξασφαλίζουν και την αξιοπρέπεια του λαού του. Θα πρέπει το δικαίωμα των κρατών να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά, να τύχει εγγύηση και οι δημόσιε υπηρεσίε πρέπει να αποκλειστούν πλήρω από την ΤΙΣΑ. Το κεφάλαιο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε πρέπει επίση να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει στι αναπτυσσόμενε χώρε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το κεφάλαιο αυτό δεν θα οδηγήσει σε αστάθεια και ταχύε διακυμάνσει των τιμών και δεν θα υποσκάψει τη βιωσιμότητα του κρατικού χρέου των χωρών αυτών. Ελπίζω ότι μετά από τη διαπραγμάτευση αυτών των συμβαστικών τροπολογιών όλοι θα υποστηρίξετε την κοινή θέση στην αυριανή ψηφοφορία ώστε να υπάρξει ένα ομόφωνο μήνυμα από την Επιτροπή ε, ανάπτυξης που θα υποστηρίξει την τελική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λόλα. Πρωτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να σας υπενθυμίσω ότι είναι εδώ παρόντες φοιτητές από τη Νέα Καλλιδονία που έχουν προσκληθεί από τον κύριο Μόρις Πόγκα για να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες της Επιτροπής μας. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Νόρμπερτ Νόιζερ, ο οποίος είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Ο σκιώδης μας συγητής δεν είναι παρόν. Γι' αυτό θα ήθελα να χαιρετήσω από τη δική μου πλευρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα αυτής της ε, διαπραγμάτευσης και την ικανοποίησή μας με την τελική γνωμοδότηση για την ΤΙΖΑ. Νομίζουμε ότι αυτή η γνωμοδότηση θα στείλει ένα στεναρό μήνυμα προς όλους τους ε, συναδέλφους μας στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και θα διευκρινίσει το γεγονός ότι ο αντίκτυπος της συμφωνίας ΤΙΣΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και επομένως θα πρέπει να υπάρξουν οι έρευνες αντικτύπου από την πλευρά της Κομισιόν για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό είναι θεμελιώδες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι συνεκτική η πολιτική μας και θα τηρηθούν οι σχετικές αρχές. Ζητούμε από την Κομισιόν να συνεχίσει να αυξάνει την ε, <clears throat> διαφάνεια και την δημοκρατική λογοδοσία στα θέματα αυτά και επίσης να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση, μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν τις διαπραγματεύσεις. Γιατί όλα αυτά τα θέματα που συζητούνται εμπλέκουν και την κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η πλήρης πληροφόρησή τους. Η δυνατότητα λοιπόν οι χώρες να αναπτύξει να συμμετάσχουν σε αυτή τη συμφωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευέλικτη προσέγγιση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ισοδίκια πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά υπηρεσιών. Σε ένα πολυμερές πλαίσιο δεν μπορούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο όπως οι αναπτυγμένες χώρες. Εξ ονόματος της μας λοιπόν Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία και ιδίως την κυρία Σάντσεφ για την πολύ καλή εργασία της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει Η Χάιντι το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η συνάδελφος ε, Λόλα Σάντσες έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά έχουμε δύο σημεία που μας προβληματίζουν. Υπάρχουν δύο τροπολογίες, ε, οι οποίες είναι ε, ουσιαστικής σημασίας. Η τροπολογία 20, η οποία λέει ότι όταν ε, θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις εκτός ε, της ε, διαδικασίας αντόχα, ενδεχομένως αυτό θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα σε αναπτυσσόμενες χώρες και το διεθνές εμπορικό σύστημα, γιατί οι επενδύσεις και τα πνευματικά δικαιώματα είναι απολύτως διασυνδεδεμένα και επομένως θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη. Και έπειτα έχουμε και την τροπολογία 22 όπου αναφέρεται ότι η συμφωνία της ενδεχομένως θα προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά στο δικαίωμα πρόσβασης ε, στην ε, τροφή ε, την, ότι γίνεται μία προσπάθεια και υπάρχει μία τάση ιδιωτικοποίησης ας πούμε της πρόσβασης στο πόσιμο νερό και τα λοιπά και ότι και αυτό το σημείο εμέσως ε, δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά τη διατήρηση των υδάτων πόρων αλλά ε, και την ε, πρόσβαση στην τροφή αλλά και στις ζωοτροφές πράγμα που με τη σειρά του δημιουργεί κίνδυνο. Τροπολογίες 20 λοιπόν και 22 μας δημιουργούν πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφός μου ο Μπέρντ Λούκερ, ο οποίος είναι σκιώδη συγητής, θέλει να ευχαριστήσει την συγγήτρια. Εμείς χαιρετίζουμε την Τίζα ως την πιο σημαντική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που έχει διαπραγματευτεί ποτέ. Είναι 23 μέλη του ΠΟΕ που συμμετέχουν και είναι πάρα πολύ νευραλγική για την φιλελευθερωποίηση της διεθνούς, του διεθνούς ε, το, μάλλον του διεθνούς εμπορίου για τις υπηρεσίες και θα οδηγήσει σε οικονομική βελτίωση για όλες τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Οι συμβασικές τροπολογίες όμως μας φαίνονται προβληματικού χαρακτήρα και δεν είμαστε σε θέση να τις υποστηρίξουμε. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη συμβασική τροπολογία 1, η οποία ζητεί από την Κομισιόν σε όλες τις ε, συμφωνίες να εξασφαλίσει την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, ορισμένα άλλα θέματα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασκήσει την ήπια δύναμή της σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί <coughs> ότι θα μπορέσει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος ή κοινωνικά πρότυπα ή πρότυπα στα ανθρώπινα δικαιώματα που να συνάδουν με αυτά των αναπτυγμένων χωρών. Όλα αυτά πρέπει να, να τα αντιληφθούμε υπό το πρίσμα της οικονομικής ανάπτυξης. Μόνο οι αναπτυγμένες χώρες μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να είναι στοιχεία των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των αμπλεκομένων ε, χωρών. Μόνο έτσι μπορούμε να οδηγήσουμε σε μια πραγματική ανάπτυξη σε ένα πιο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο λοιπόν αυτές οι δεσμεύσεις και όχι να θεωρηθούν προαπαιτούμενα. Επίση, στην τροπολογία υπαριθμών δύο συνδεσμού ζητάει η Κομισιόν να υπάρξει βελτίωση της ε, αντιμετώπισης της κοινωνίας των πολιτών και των εργατικών συνδικάτων. Αλλά η διαπραγμάτευση αυτή δεν γίνεται εν γέννη στο δημόσιο τομέα. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν έχει καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και στην πραγματικότητα είναι υποδειγματική η διαφάνεια στα θέματα της διαπραγματεύσης της ΤΙΖΑ γιατί η Κομισιόν κάνει ε, σαφή και τακτική πληροφόρηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διοργανώνει ε, διαβουλεύσεις με εμπλεκόμενους φορείς και με την κοινωνία των πολιτών έχει λοιπόν εκπληρώσει την ανάγκη της ε, διαφάνειας. Τροπολογία 4. Ζητά να υπάρξει μια συμφωνία που γίνεται δεκτή από όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Δυστυχώς είναι περιορισμένος ο αριθμός των χωρών υπό ανάπτυξη που συμμετέχουν στη συμφωνία αυτή. Αυτή η δομή της ΤΙΖΑ όμως θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του ΠΟΕ και το, η φιλελευθερωποίηση της ε, εμπορίας υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται ανοιχτή σε όλου. Η Κίνα είναι μια από τι χώρε οι οποίε έχουν τονίσει ότι θέλουν να εμπλακούν σε μια τέτοια συμφωνία. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στου διαπραγματευόμενου από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κίνητρα ώστε να μπορέσουν και άλλε χώρε να υποστηρίξουν του στόχου τη ε, ΤΙΖΑ. Και έρχομαι τώρα στο, στην τροπολογία 7 για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Παραδείγματο χάρη πρόσβαση σε πιστώσει. Όλα αυτά μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, ανάπτυξη μιας χώρας. Αλλά δεν μπορούμε για το λόγο αυτό να δεχτούμε αυτά που περιέχει η συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία είναι πολύ περιοριστική. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω ως σκιώδης του ΕΛΚ για αυτή τη χνομοδότηση. Ευχαριστώ τη Λόλα για τη δουλειά της και τους άλλους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες, τους άλλους κοιόδης, γιατί συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Αν και αρχίσαμε από διαφορετικά σημεία κίνησης, καταλήξαμε πολλές φορές σε συμβιβασμού ιδίως για τα θέματα της ανάπτυξης, που αυτό είναι το θέμα που θέλουμε να τονίσουμε στην χρηματοδότησή μας για την ΤΙΣΑ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω από απόψεως ΕΛΚ δύο συμβιβαστικές όπου που πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ελπίζουμε η αρμόδια καθήλυνη επιτροπή να το λάβει υπόψη της επιτροπή τα δηλαδή. Γιατί δηλώνουμε ρητά ότι οι υπηρεσίες και το εμπόριο υποζημισμένες συνθήκες βέβαια μπορούν να είναι μοχλός για βιώσιμη ανάπτυξη, μείωση της ανέχειας και των ανισοτήτων καθώς και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται λοιπόν για διατύπωση που τονίζει ιδιαίτερα το αναπτυξιακό. Είναι σημαντικό μήνυμα δηλαδή που στέλνουμε από την Επιτροπή μας. Καθώς και η διατύπωση που δεχτήκαμε στην συμβιβαστική 4 δηλαδή την απόρριψη οποιασδήποτε ρήτρας που θα ήταν ασύμβατη με το ΓΑΤ ε, πρέπει η ΤΙΣΑ νομίζουμε να παραμείνει ανοιχτή για τις αναπτυσσόμενες χώρες ανοιχτή. Και οι άλλοι ισχυώδεις από τις άλλες πολιτικές ομάδες τα ίδια είπαν. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και άλλα θέματα που, που δεν μας αρέσουν και τόσο, αλλά για να επιδείξουμε συμβιβαστικό πνεύμα καταφέραμε να τα εξισορροπήσουμε όλα. Συγχαίρω λοιπόν ξανά τη Λόλα. Αυτά από μένα. Τώρα η Καμισιόν. Κυρία Γκίντερακ Κέμικ Κλίνερ. Χαίρετε. Γκίντερακ και Μακίνα από τη Γενική Εμπορίου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την γνωμοδότηση, την οποία διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή ε, καθώς και τις ε, τροπολογίες ε, όσον αφορά την διαφάνεια διαπιστώνω ότι πολλές προσπάθειες έχουν γίνει έτσι ώστε ε, ε, όλα τα έγγραφα της ε, διαπραγμάτευσης να είναι διαθέσιμα. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τώρα την αρχιτεκτονική της συμφωνημένης διαπραγμάτευσης, διαπραγμάτευσης που ήδη αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα στη Γενέβη. Είναι, είναι προφανές ότι ευθυγραμμίζεται με την αρχιτεκτονική ε, της, ε, των συμφωνιών ΓΚΑΤ και των διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και είναι ανοιχτές ε, στις χώρες όλες και περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία και εσείς υπογραμμίσατε εδώ. Δεν νομίζω ότι έχω λόγο να πω κάτι άλλο. Δεν υπήρξαν συγκεκριμένε ερωτήσεις, επομένως αυτά ήθελα να πω και σα ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα τώρα να ξαναγυρίσω στην Λόλα για να μας δώσει τα τελευταία της συμπεράσματα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους σκιώδης ε, εισηγητής. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως ε, οι περισσότερες ε, ομάδες έχουμε δώσει έτσι κάποιες, έχουμε κάνει κάποιες υποχωρήσεις και νομίζω ότι όλοι έχουμε στηρίξει και τις κόκκινες γραμμές μας. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Αυτά και σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε αύριο για αυτήν την το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά ή να αρχίσουμε απευθείας. Είναι ήδη οι ομιλητές εδώ. Νομίζετε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το επόμενο θέμα λοιπόν είναι η ε, κοινή συνεδρίασή μας με την Υποεπιτροπή ε, Ασφάλειας και Άμυνας ΣΕΝΤΕ και επομένως μπορώ να καλέσω τους ε, ομιλητές έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την διαδικασία. Παρακαλώ.